Sorry. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε τώρα. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε. Θα συνεχίσω στη γλώσσα του Δάντη. Αλλά καθίστε στα αγγλικά και βλέπουμε. Λοιπόν, φάλατε τα ακουστικά σας. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Καταρχήν σας καλωσορίζω όλους και όλες. Είναι σήμερα η πρώτη μας συνεδρίαση αυτής της θητείας. Ελπίζω λοιπόν η συνεργασία μας να αποβεί θετική και ωφέλιμη. Προτείνω πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη που έχει δύο σημεία και τα δύο αφορούν την αξιο... τον προϋπολογισμό όπως ήταν γνωστό από πριν λοιπόν, Θα εξετάσουμε τα δύο σημεία μαζί. Έχουμε και αναμετάδοση, να το ξέρετε, στο ίντρανετ. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις. Υπάρχει πολιτική συνένεση στη διάσκεψη των Προέδρων δηλαδή, των Επιτροπών, καθώς και συμφωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Γιούνκερ, να γίνουν νωρίτερα οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να οργανώσει τις ακροάσεις αυτές έγκαιρα ώστε να μπορεί να γνωμοδοτήσει και να μπορέσει έτσι η νέα Επιτροπή Κομισιόν να αρχίσει τις εργασίες της από την 1η Νοεμβρίου. Επομένως, θα χρειαστεί να οργανώσουμε μια έκτακτη συνεδρίασή μας, τουλάχιστον μία, τον Σεπτέμβριο ήδη, για τους ε, υποψήφιους επιτρόπους που αφορούν τα θέματά μας. Την πρώτη εβδομάδα μετά το Στρασβούργο του Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό Τη πρώτη ακρόαση. Βέβαια οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί αλλά οπωσδήποτε ήθελα να το ξέρετε από τώρα για να το λάβετε υπόψη στο πρόγραμμά σας. Δεύτερον, αυτή ήταν για την έκτακτη συνεδρίασή μας. Δεύτερον, μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία το 7ο βραβείο Λούξ να σας πω περί τίνος πρόκειται. Από το 2007 το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί ένα βραβείο σε κάποιο κινηματογραφικό έργο ευρωπαϊκό ή συμπαραγωγή. Είναι το μοναδικό τέτοιο βραβείο που χορηγεί κοινοβούλιο. Είναι το βραβείο Λουξ λοιπόν. Γενικά χορηγείται σε ένα έργο, σε μια παραγωγή που αφορά θέμα που ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο και την Ευρώπη. Είναι μια πολύ θετική χειρονομία προς την κινηματογραφική βιομηχανία της Ευρώπης και αφορά ιδίως απευθύνεται σε νέους σκηνοθέτες. Έχουν επιλεγεί 8 έργα φέτος, ε, μάλλον και αν, έχετε αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες το Κάρλο Βιβάρη αποφασίστηκε αυτό κοιτάξτε στο ίντερνετ Lux Prize θα γίνει πάντως διάσκεψη τύπου σήμερα στη Ρώμη για την έναρξη, επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Βενετίας αρχίζει βέβαια 27 Αυγούστου και θα ανακοινωθούν di Venezia durante le giornate ε, Τρία βραβεία. Οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και εγώ έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε και θα παρουσιαστούν οι τρεις υποψηφιότητες στις 24 γλώσσες της Ένωσης. Λοιπόν, θα μάθουμε λοιπόν τότε τα τρία ονόματα και θα σας δώσουμε τα τρία ονόματα που θα επιλεγούν για το βραβείο Λουξ. Και θα σας δώσουμε τότε περισσότερες πληροφορίες. Ο κάθε βουλευτής αν θέλει μπορεί να δει αυτά τα έργα και να επιλέξει εκείνο που του αρέσει περισσότερο για το βραβείο Λουξ 2014. Θα τα ξαναπούμε όμως τον Οκτώβριο στην τακτική μας συνεδρίαση. Αν δεν έχει κανείς κανένα σχόλιο, α, ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλού νέους συναδέλφους. Δεν έχει μικρόφωνο η μιλήτρια και δεν ακούγεται όμως. Um, yes, so... Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω το εξή. Έχουμε πολλούς νεοεκλογέντες συναδέλφου. Συγχαρητήρια. Να του πω ότι ε, αυτό το έπαθλο, αυτό το, το βραβείο Λούξ είναι μια ιστορία πετυχημένη εδώ για το Κοινοβούλιο. Μεγάλη επιτυχία. Ε, δείχνει το ότι είμαστε προσιλωμένοι στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όλοι οι νέοι συνάδελφοι να λάβουν μέρος, να βοηθήσουν στην επιλογή, να τα προωθήσετε στην εκλογική σας ε, περιφέρεια, γιατί αυτό είναι τμήμα της ε, επικοινωνίας σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσετε την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρόεδρος. έργασε ευχαριστούμε. Βεβαίως και πολύ καλύτερα θα τα συζητήσουμε τον Οκτώβριο του βραβείου Λουξ και να συμμετάσχουμε βεβαίω. Τίποτα άλλο για αυτό το θέμα τώρα, αν δεν ζητεί άλλο το λόγο, οπότε πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση 2015. Και πιο συγκεκριμένα βέβαια έχουμε τις σχετικές παρατηρήσεις όπως προβλέπει η διαδικασία. Όπως εσείς γνωρίζετε, σας υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή τέλη Απριλίου παρουσιάζει τον προπολογισμό. Φέτος, βέβαια, οι σχετικές εκτιμήσεις έγιναν στις 11 έκτου, ξέρετε για ποιον λόγο, λόγο της προεκλογικής εκστρατείας και το σχέδιο προϋπολογισμού για τη χρήση 2015 ε, η παρουσίαση 25 Ιουνίου. Τότε είναι, οπότε και ακολούθησαν οι ανταλλαγές απόψεων. Οπότε είχαμε υστέρηση δύο μηνών για αυτή την δημοσιοποίηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού λόγω των εκλογών και ελπίζω να έχουν περισσότερο χρόνο από του χρόνου. Και βέβαια όλα αυτά, σαν διαδικασία, ισχύουν για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τώρα, τι κάνουμε. Πρώτον, πρέπει να εγκρίνουμε το κείμενο με μια γνωμοδότηση που ε, ορίζει τις προτεραιότητες της δικής μας επιτροπής. Δεύτερον, θα πρέπει να εγκρίνουμε κάποιες τροπολογίες που αφορούν τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά του συγκεκριμένου ε, σχεδίου προϋπολογισμού. Και εγώ συντάκτηρα έχω την υποχρέωση της παρουσίασης αυτής της γνωμοδότησης. Υπάρχει πίεση χρόνου γιατί θα πρέπει η γνωμοδότηση να εγκριθεί και θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο συγκεκριμένη έκταση, συγκεκριμένο όγκο αυτή η γνωμοδότηση 200 λέξεις και οπότε έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες και δικές μου σήμερα πάνε εκεί που θα πρέπει να τις εγκρίνουμε τώρα όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία εμείς θα θέλουμε να τροποποιήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Όμως, μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία όσον αφορά την θέση του Συμβουλίου. Θα προκύψει κάποια στιγμή, ενώ ακόμα συζητούμε τις τροπολογίες, οπότε ε, αφορούν οι τροπολογίες μας στο σχέδιο μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τροπολογούμε τώρα με αυτές τις Και τελούμε εν αναμονή της θέσης του Συμβουλίου. γενικώ το Συμβούλιο προβαίνει σε κάποιες περικοπές. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θέση θα υιοθήσει στο το Συμβούλιο στο τέλος Αυγούστου. Και υπάρχουν βέβαια φήμες ανεπίσημες, ότι δηλαδή έχει συμφωνήσει για το συνολικό ποσό κάθε τίτλου και ξέρουμε για τον τίτλο, τρίτο, τίτλο, τρίτο κεφάλαιο του προπολισμού, εκεί που έχουμε το Ευρώπα Κρεατίβα, Ευρώπη των Πολιτών και την επικοινωνία, εκεί υπάρχει περικοπή 3,3% που είναι προγράμματα που ενδιαφέρουν τη δική μας Επιτροπή. Και έχουμε πέρα από αυτά άλλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν υποστεί σημαντική μείωση όπως το Erasmus Plus. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα πει η Επιτροπή και αυτή η περικοπή θα πρέπει να μελετηθεί μέχρι πού θα φτάσει ούτως ώστε να μην θίξει αυτά τα πολιετή προγράμματα. Πρόκειται για, άλλωστε για, την, για το πρώτο έτος της, του επταετούς προγραμματισμού της ΛΕΣ του Κοινοβουλίου. Θέλω να υπάρχει πως μια εγκάρσια, ε, μια εγκάρσια εντολή, το ώστε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα ποσά εκεί όπου το Συμβούλιο έχει επιφέρει αυτές τις περικοπές. Οπότε μπορούμε να προτάξουμε αυτές μας τις τροπολογίες όσον αφορά τη γνωμόδοτηση και όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά. Τώρα, θα πρέπει να γίνει επομένως η ψηφορία σε σχέση με αυτή την εγκάρσια η οριζόντια εντολή, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ε, αν θέλετε ψηφίζουμε με ανάταση, χειρός. Συμφωνείτε, ναι, ωραία. Επίσης, είναι δυνατόν μετά να συζητήσουμε τα του δικού μου κειμένου. Έχουμε τα, αυτά τα πολιτικά προγράμματα, αφορούν μια αιτία, ε, για εκπαίδευση, κατάρτιση, αθλητισμό, τα, τα μέσα ενημέρωσης στους πολίτες λοιπά. Αυτή είναι η τίτλη των σχετικών προγραμμάτων, οπότε τώρα Έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία κλείσαν την πρώτη χρονιά την μπαίνουν στη δεύτερη και επομένω είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα του στόχου κάθε προγράμματο και να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει σχέση με τη στατική 2020. Πρόκειται για μια διαβούλευση. Τώρα η οποία βρίσκεται εν εξέλιξη, είδε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα προβεί σε κάποια αναθεώρηση των προτάσεών τη Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Και έχουμε και το Erasmus Plus, εκεί που υπάρχει μια σημαντική αύξηση της πρικοδότησης. Στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Ε, quindi noi Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει έτσι και αλλιώς να δούμε το πώς θα πετύχουν τους στόχους μας. Αυτό έχει σημασία και όσον αφορά τις πιστώσεις των πληρωμών αλλά και τις πιστώσεις υποχρεώσεων στα διπλαίσια του Erasmus Plus έχουμε μια σειρά ή υποπρογραμμάτων το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως όπως το Λεωνάρντο και άλλα όλο ένα και περισσότερο επιβάλλεται να υπάρχει περισσότερη κινητικότητα και διδασκόντων και φοιτητών Γι' αυτό και πρόκειται εδώ για ακόμα μια σημαντική επιτυχία. Επομένως χρειάζεται επαρκής προοικοδότηση και πιστός πληρωμών, τόσο ώστε να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Το 2012 με μια τροπολογία μας πετύχαμε την αύξηση της σχετικής προϋποδότησης με πιστώσεις πληρωμών για το Erasmus Plus. Επομένως εδώ έχουμε διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο γιατί είναι πάρα πολύ δημοφιλές το, το έρασμος ε, στους νέους στην Ευρώπη. Άρα μεγάλη προσοχή και έτσι να μην καταρρεύσουν οι πιστώσεις για το έρασμος. Επίσης κάτι άλλο που να προβληματίζει είναι το πρόγραμμα Μαρή Curie το οποίο αφορά τους νέους ερευνητές. Έχει να κάνει και με την δουλειά της δικής Επιτροπής και βεβαίως και αφορά τους νέους ερευνητές και το πρόγραμμα της πολιτικής ενόψης του 2020 και επίση εδώ σημαντικό το προτινόμενο δίκτυο το οποίο θα αποτελέσει το μέσο διαχείρισης της ψηφιακής κληρονομιάς. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε να μην επιβληθούν περικοπές. Θα πρέπει να προσχεθούν εξηγήσει για ό,τι προτείνουν. Δημιουργική Ευρώπη ήταν ένα άλλο πρόγραμμα το, για το οποίο ήμουν υπεύθυνη την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία. Εδώ προβλέπεται για τις πιστώσεις ε, υποχρεώσεων μία μικρή περικοπή. Και για την Δημιουργική Ευρώπη είχε προβλεφθεί μία αύξηση 9%. Θα πρέπει σε όλα αυτά τα μέτωπα παραλλήλως να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να μας παρασχεθούν εξηγήσει και φαντάζομαι ότι οι σχετικές περικοπές πρόκειται να αιτιολογηθούν πρώτα-πρώτα από το ότι έχουμε κάποια μεταφορά των ε, κονδυλίων εγγύησης προς τη χρήση 2016 και από την άλλη μεριά άλλη μια αιτιολόγηση είναι ότι η χρηματοδότηση αυτών των πολιτών προγραμμάτων πρόκειται στο μέλλον να αυξηθεί. Εν πάση περιπτώσει πρόκειται να μας εξηγήσει η Κομισιόν γιατί προτείνει αυτά που προτείνει που αφορούν τόσο πολύ την πολιτική μας εδώ. Τις δεσμεύσεις μας. Οπότε βέβαια να μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί και άλλα προγράμματα όπως την πολιτική πρωτεύουσα το πολιτιστικό παρατηρητήριο και επομένως βλέπετε ότι έχουμε προγράμματα και υποπρογράμματα. Μιλούμε για τον τρίτο τίτλο, τρίτο κεφάλαιο του προπολογισμού. Εκεί υπάγεται αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει επομένω να τοποθετηθούμε σε όλα αυτά και εγώ ως εισηγήτρια πρόκειται να έρθω σε επαφή με άλλες πολιτικές ομάδες και να ε, παρουσιάσω συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά και αυτό το τρίτο κεφάλαιο. Ε, θυμάμαι μία μακρά συζήτηση σε σχέση με την Επιτροπή τη δική μας, σε σχέση με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο που είχαμε κάνει, που τελικά όμως θα έπρεπε να υποστούμε μια μεγάλη περικοπή τότε είχαμε περικοπή του προπολογισμού το 2013 κατά 20% και θυμάμαι ήταν η συνάδελφος Τάκουλα ε, η εξαιρετική μας ε, εισηγήτρια τότε αφορούσε σχολεία, τους ευρωπαϊκούς πολίτες, ε, νομικά πρόσωπα ενώσεις πολιτών και είπαμε ότι θα πρέπει σωστές πρωτοβουλίες επικοινωνίας να προβάλλουμε κάποια προγράμματα που αφορούν 15 χώρες, αφορούν το ραδιόφωνο και έτσι θα υποστηρίξουμε την επικοινωνία στην Ευρώπη σε αυτά τα θέματα. Μιλούμε για 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ακούν ραδιόφωνο ε, για τέτοια πολιτικά θέματα. Οπότε εκεί να πέσει αυτή, αυτό το, το ψαλίδι είναι κρίμα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να εξηγήσουμε τις προτεραιότητες μας. Τώρα θα δώσω τον λόγο εις όποιον το έχει ζητήσει. Ε, και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί που όλων αυτών. Οι συνάδελφοι έχουν τον λόγο πρώτα. Κριστίνα, κατόπιν η κυρία Τρούπελ στα πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε γιατί η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ που τονίσατε ιδιαίτερα τα σημεία που θα είναι η βάση της γνωμοδότησής μας. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο αλλαγές. Πρώτον για το σημείο 2 σε ορισμένες χώρες μέλη γίνονται προσπάθειες επιβολής ενός ειδικού φόρου για το έρασμος 2 συν. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω εδώ μια φράση που να λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να φορολογούνται για τον έρασμο 2. Και κάτι άλλο ακόμα. Θα ήθελα να σκεφτούμε μήπως δεν θα έπρεπε να προσθεθεί ένα σημείο 6 όπου να ζητούμε από την Κομισιόν πληροφόρηση για την κατανομή των δαπανών αναπρόγραμμα στις διάφορες χώρες μέλη για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια για ως προς την δαπάνηση του δημοσίου χρήματος. Θα καταθέσω λοιπόν αυτές τις δύο τροπολογίες γραπτός. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιμπέτσκα. Τώρα η Χέλγα Τρούπελ. Και εμείς οι πράσινοι είμαστε αντίθετοι με τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο. Μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα Greater Europe. Σημαντικό για την δημιουργία της πολιτιστικής πολυμορφίας μέσα στην Ευρώπη. Είμαστε κατά λοιπόν των περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο, γι' αυτό θα επαναφέρουμε τα αρχικά νούμερα που προβλέπει ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θέλουμε και Euronet Plus να μπορούν να λειτουργήσουν. Πρόκειται για ραδιοφωνικούς σταθμούς που επιθυμούμε να μπορούν να μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά μηνύματα. Και πάνω σε αυτά θα εργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Μίτσι. Είμαι νέα Ευρωβουλευτής. Καλημέρα. Ορισμένα πράγματα βέβαια δεν θα τα γνωρίζω, μιας και δεν ήμουν βουλευτής πιο πριν. Το γραφείο μας στη Μάλτα εντοπίζει ένα πρόγραμμα Share Europe Online δηλαδή η Ευρώπη επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Φαίνεται πως οι βουλευτές οι οποίοι υποστήριζαν το πρόγραμμα αυτό ή ο βουλευτής ή η βουλευτής δεν ξέρω δεν είναι πια στην Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων. Γι' αυτό και ρωτά το γραφείο μας τι, κάνει, τι γίνεται με το πρόγραμμα Europe Online, αν έχει υποστεί περικοπές ο προπολογισμό του. Και το δεύτερο, μια και εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων, να έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας, να έχουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Τα Μαλτέζικα αποσιάζουν σήμερα. Καταλαβαίνω κύριε Μίτση και τώρα. Κύριος Ντρογεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θέλω να σας παρουσιάσω έναν άλλο προβληματισμό. Όλοι βρεθήκαμε στην περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο και είδαμε την φοβερή τραγωδία στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι πρέπει να εκφράσουμε άποψη. Μία από τις τροπολογίες αναφέρεται στο πρόγραμμα της Ανατολικής Γειτονίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προβλέπει και συνεργασία βεβαίως και σε πολιτιστική συνεργασία. Και ιδίως για τους νέους ανθρώπους στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τις προτεραιότητες αυτές. Είναι θεμελιώδες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που είναι αρμόδια όπως εμείς για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κτλ. να στραφεί ιδίω προς τους νέους. Γιατί έτσι θα ανοίξουμε τον δρόμο για την ενίσχυση της ανεκτικότητας της πολιτιστικής συνεργασίας και έτσι μπορούμε να εργαστούμε ορθολογικά, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε, να βάλουμε τις βάσεις για μια συνεργασία στο μέλλον και ιδίως μια εταιρική σχέση με μια γενιά η οποία θα διαδραματίσει κέριο ρόλο στο μέλλον μας. Βέβαια, λόγω των ευρωεκλογών, των πρόσφατων ευρωεκλογών, φέτος έχουμε λίγο χρόνο για την συζήτηση του προπολογισμού. Άλλε φορέ ήταν είναι διαφορετικά. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει ωστόσο σε βάθος. Να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τη και να μας επιτρέπει να πάμε σε βάθος. Γιατί ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμό είναι σημαντικά πράγματα για την νεολαία και χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Άλλωστε, είναι σημαντική και η χρηματοδότηση που προβλέπουν οι χώρες μέλη στους δικούς τους εθνικούς προϋπολογισμούς για τα θέματα αυτά. Εγώ έχω υποβάλει τρεις τροπολογίες, το περιεχόμενο των οποίων ξαναβρίσκω και σε άλλες τροπολογίες που έχει υποβάλει και η Πρόεδρος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θέματα αυτά μπορούν να πετύχουν ευρεία συνένεση εδώ για παράδειγμα ΕυρωΝΕΤ, εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Euronet είναι η συνεργασία των διαφόρων ραδιοφωνικών σταθμών. Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα των ενδεχόμενων περικοπών στη χρηματοδότησή τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις περικοπές αυτές, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί και στο μέλλον η εργασία τους διότι αν απειλείται ο προϋπολογισμός τους υπάρχει μέγα θέμα. Υπάρχουν και τα προγράμματα για τον αθλητισμό. Εδώ τίθενται θέματα όπως ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και εδώ πρέπει να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα οργανώσεις, που προωθούν τον αθλητισμό για λόγους υγείας του πληθυσμού, αλλά και για την είσοδο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μίλησαν και για την τραγωδία στην Ουκρανία, που κατά τη γνώμη μου η αντίδρασή μας πρέπει να εντάσσεται μέσα στην ανατολική γειτονία. Εκεί όμως ο προϋπολογισμός μας είναι πολύ περιορισμένος, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι και τη συνεργασία μας με τους νέους και να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός εκείνος χώρος που θα αποτελέσει το θεμέλιο για να αποφευθούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον. Έχω και λίγες παρατηρήσεις τώρα για 10-12 ακόμη τροπολογίες. Έχω και μια παράκληση προς την Πρόεδρο. Τα προγράμματα που φτάνουν στη λήξη τους και που είναι δέκα περίπου και που σύντομα πρόκειται να λήξουν. Να τους δοθούν νέες καλύτερες προοπτικές. Να δούμε τα προγράμματα αυτά ποια αποτελέσματα επέτυχαν και ποια μπορούν να είναι τα νέα στοιχεία τα οποία θα μπορούν ή τα νέα προγράμματα τα οποία θα επιτρέψουν τη συνέχιση των προσπάθειών αυτών χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Οι υφιστάμενε γραφειοκρατικέ διαδικασίε πρέπει να διαμορφωθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ότι ορισμένε χώρε μέλη διαθέτουν ιδίους πόρου το πρόγραμμα Ευρωπεάνουμ έχει επαρκή προϋπολογισμό, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα Έχει αρχίσει ικανοποιητικά βέβαια, έχει χρηματοδότηση από τις χώρες μέλη, αλλά δεν είναι βέβαιο το μέλλον του. Για το έρασμος τώρα, θα επανέλθω στα όσα είπε η συνάδελφός μου κυρία Βιβάτσκα προηγουμένως, δεν θα προσθέσω τίποτα, αλλά θέλω να επισημάνω ένα πράγμα. Το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτά εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Γίνονται προσπάθειες που είναι όμως κατακαιρματισμένες και δεν συνδέονται καλά μεταξύ τους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την βία κατά των δημοσιογράφων, θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή του δικαίου, αλλά δεν έχουμε πάντα τις αρμοδιότητες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα. Κυρίω πρόκειται για την εκπαίδευση των μέσων αλλά και διά των μέσων, με τη βοήθεια δηλαδή των μέσων ενημέρωσης. Αυτή η εκπαίδευση χρειάζεται οπωσδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να θυμηθούμε ιδίω βέβαια τα θύματα της Αεροπορική τραγωδίας. Δυστυχώ λινθμόνησα να το κάνω στην αρχή. Η σκέψη μας είναι διαρκώς στα θύματα και στις οικογένειές τους. Για τα θέματα τώρα <clears throat> που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά όπως εξηγήσατε πρέπει να έρθουμε σε διάλογο και με άλλες χώρες. Ναι, εσείς παρακαλώ κυρία μου. Κοιτάξτε, ως νέα ευρωβουλευτής ε, τελώ εν συγχύση, το ομολογώ με όλα αυτά που ακούω. Και διαρωτώ με, δεν μάθαμε τίποτα από τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ξοδεύουμε εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για να προωθούμε μια προπαγάνδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τόσα εκατομμύρια εκλογής απέρριψαν το, ευρωπαϊκό, το έργο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η εκλογική μου περιφέρεια θα φρίξει αν δει τις δαπάνες αυτής της Επιτροπής. 60 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται για να φτιαχτεί ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ενώ εκεί αναγκάζονται να κάνουν τράπεζες τροφίμων για να ζήσουν τις οικογένειές τους άλλα εκατομμύρια δίνονται για ανταλλαγέ σπουδαστών. Ενώ πρέπει να βοηθήσουμε εκατομμύρια νέους που είναι άνεργοι και που δεν έχουν ούτε εκπαίδευση. Πρόκειται για μια εσχρή δαπάνη των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Οι άνθρωποι χρειάζονται πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και αυτή η κατασπατάληση του χρήματος προσπαθώντας να αρπάξετε από εδώ και από εκεί ό,τι μπορείτε, είναι ακριβώς αυτό. Κατασπατάληση. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ περικοπής παντός κονδυλίου της Επιτροπής Πολιτιστικών. Έχω πραγματικά φρίξει με αυτά που ακούω εδώ. Καιρός είναι να ακούσετε τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι λαοί της Ευρώπης. Ναι, κύριε Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πλατφόρμα στην οποία θα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνένεση σε σχέση με το τι ωφελεί όλο τον κόσμο. Έχουμε εδώ πέρα πολύ, πολύ συλλεκτικότητα απόψεων και θεμάτων. κοιτάξτε, αυτά που μόλις άκουσα με αφήνουν άφωνοι. Ειδικά όταν ακούει κανείς τους ανθρώπους τι λένε οι πολίτες ακριβώς αυτά τα πράγματα τους ενδιαφέρουν. Η προώθηση του πολιτισμού, τα προγράμματα ανταλλαγής ενδιαφέρουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτά που οδηγούν σε μια ευρωπαϊκή συνύπαρξη. Και αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι μια ένωση, τότε τα προγράμματα αυτά είναι απαραίτητα. Εμείς δεν ασχολούμαστε μονάχα με τις γερμανικές περιφέρειες, μέσω των συνεργασιών με άλλες πόλεις, της ανταλλαγής πολιτιστικών προγραμμάτων, φτάνουμε και γνωρίζουμε τους άλλους πολιτισμούς δεν ασχολούμαστε μόνο με την πατρίδα μας και, και το κόμμα UKIP της Μεγάλης Βρετανίας ας ανοίξει τα μάτια του, ας κοιτάξει τι γίνεται και σε άλλες χώρες και ίσως αυτό να τους βοηθήσει να ανοίξουν και το πνεύμα τους. Χαίρομαι που στον τομέα του πολιτισμού λαμβάνουμε και από τις χώρες μέλη σαφή αύξηση των ε, ε, χρηματοδοτήσεων για το Εράσμους συν μας προσφέρουν περισσότερα χρήματα, ειδικά για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα ανταλλαγών. Ωστόσο, κινδυνεύουμε και εδώ από περικοπέ. Εμείς θα θέλαμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός τους, διότι αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει τόσο μεγάλη αξία για τους ανθρώπους, όπου οι άνθρωποι με αυτές τις άμεσες ανταλλαγές έχουν γνωρίσει η μεν τους δε. Εδώ πρέπει και τα γραφειοκρατικά κατόφλια να μειωθούν και ο προϋπολογισμός να αυξηθεί. Και αυτός είναι ο ρόλος μας της Επιτροπής Πολιτισμού. Και εφόσον καλούμαστε να δαπανίσουμε για τα πράγματα αυτά χρήματα των φορολογουμένων, ε, κάνουμε. Είναι άξιος ο σκοπός αυτός, αποδίδει γιατί υπάρχουν και άλλες δαπάνες όπως αυτές για παράδειγμα για την αγροτική οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας που μου φαίνονται πολύ λιγότερο δικαιολογημένες. Νηριάντα. Και, εγώ είμαι καινούργια βουλευτής από την Ιρλανδία και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τις πολιτιστικές προεδημιουργικές βιομηχανίες στις επενδύσεις γιατί οι παραδοσιακές βιομηχανίες βλέπουμε ότι βρίσκονται σε παρακμή ενώ οι πολιτιστικές σε αύξηση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για την καλύτερη κατανομή των επενδύσεων. Έπειτα, γνωρίζω ότι έχουμε πίεση χρόνου, αλλά μήπως μπορούμε να καθυστερήσουμε το, τη διορία κατάθεση τροπολογιών μέχρι μετά το Σαββατοκύριακο, ώστε ιδίω οι καινούργοι βουλευτές να μπορούν να τα δουν τα πράγματα λίγο πιο με περισσότερο χρόνο. Σας... Ναι, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται μια που όπως είπαμε και την τελευταία φορά αυτό είναι η ρυθμίση που αφορά όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και είναι μια γενική ρύθμιση. Ναι, είναι η αρχή, είναι λίγο πιο δύσκολα αλλά βεβαίως έχουμε προσαρρογή μας στην ε, γραμματεία του συμβούλου μας και τώρα λόγο έχει ο κύριος Τούτου Τούτ, του, πώς λέγεστε. Η Άλντε χαίρεται για το ότι εσείς αναλάβετε τον προϋπολογισμό αυτό θα αναδείξει περισσότερο την εκθεσή μας. Συμφωνούμε με τις προτεραιότητες όπως τις τονίσατε. Θα σας υποστηρίξουμε. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια οπότε και θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε τοποθετηθεί ήδη για τις τροπολογίες πρώτα πρώτα θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι δύο συνεχείς δράσεις που η άλλη έχει προτείνει για την Ευρώπη την επιγραμμική και την Ενεργή Ευρώπη, ούτω ώστε να μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα με τον κόσμο. Και οι εμπλεκόμενοι στα πολιτιστικά θα πρέπει με τον κόσμο να ε, συνεργαστούν και θα πρέπει ο κόσμος να συμμετάσχει περισσότερο. Δεύτερον, είμαστε υπέρ της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά ε, τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο ευρωπαϊκές δραστηριότητες να αγγίξουν τον κόσμο, να βρούμε τον καλύτερο τρόπο, τον πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση κόστος αποτελέσματο για αυτά τα δίκτυα. Τρίτον, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την πρικοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινηματογράφου. Και για αθλητισμό επίσης να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητε που οργανώνονται στα κράτη-μέλη και επίσης να δείξουμε στον κόσμο το πόσο καλός αθλητισμός για την ε, καθημερινή ζωή τους. Έχουμε επίσης τις δύο τροπολογίες του ΕΛΚ όσον αφορά το κέντρο μέσων ενημέρωση και δημοσιογράφων και πλουραλισμού πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά ιδρύματα που αφορά την ελευθερία του τύπου. Ε, Κυρία Τούμ, σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Λέζος. πρέπει να ευχηθούμε καταρχήν καλή αρχή στην αναρκτήρια αυτή συνεδρίαση και να ανταποκριθούμε όλοι στο περιεχόμενο του πολιτισμού και της παιδείας που έχουμε ενταχθεί. Εάν θέλουμε πραγματικά μια Ευρώπη του πολιτισμού, μια Ευρώπη που τη δόξασαν ο Γκέτε, ο Σέξπιρ, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Ρέμπραντ, ο Μπετόβεν, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Ρούμπενς, ο Σούμπερτ και πιάδα ολόκληρη δημιουργών πνευματικών ανθρώπων πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να δούμε το τι κάνουμε. Δυστυχώς εγώ δεν είχα μπροστά μου, δεν μου στάλθηκε ο προϋπολογισμός, δεν τον γνωρίζω και δεν μπορώ να ξέρω εάν αληθεύει το γεγονός ότι δίνονται κοντήλια για έργα της Κομισιόν. Λέω ένα παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να εφοδιαστούμε με όλα τα στοιχεία και αν είναι δυνατόν να απασχοληθούμε με άλλη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή καταστρέφονται τα τοπονύμια στην Κύπρο είναι διεθνώς απαράδεκτη η αλλαγή των τοπονημίων. και η Κύπρος κατέχεται έδαφος ευρωπαϊκό, κατέχεται από στρατεύματα τα οποία έχει πάρει απόφαση και το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αποσυρθούν. Νομίζω ότι πρέπει μία από τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής μας είναι η καταγγελία του γεγονότος της αλλαγής των προσωνυμίων και έχουμε και πληροφορίες για καταστροφή και εκκλησιών. Αλλά το γεγονός της αλλαγής των προσωνυμίων είναι αναμφισβήτητο. Όπως επίσης και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στο γεγονός ότι η σύγκρουση στην Παλαιστίνη αφορά και καταστροφή σχολείων. Είμαστε Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Παιδείας. Και γι' αυτό νομίζω ότι εάν μείνουμε απαθείς μέσα στην ασφάλεια που έχουμε σήμερα εδώ, εμείς είμαστε ασφαλείς και κλείνουμε τα μάτια, στρούθοκαμιλίζουμε μπροστά στα γεγονότα που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, νομίζω ότι δεν επιτελούμε το έργο μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκλέζο, κύριος Γουόρτ. Η κυρία διορθώνει πρόεδρος. Για μένα είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να παρουσιάσω μια πιο αληθινή περιγραφή του τι συμβαίνει στα βορειοδυτικά της Αγγλίας. Όταν ακούμε αυτά που λέει η Λουίς Μπρούς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εκλογέων γιατί είμαστε από την ίδια περιφέρεια. Ντρέπομαι που είμαι στην ίδια αίθουσα με κάποιον που είναι τόσο αρνητικός για τον πολιτισμό και για το μήνυμα που στέλνει αυτό στους πολίτες. Θα έπρεπε να συμμεριστούμε τα πολιτισ... τον πολιτιστικούς μας θησαυρού και να αναλάβουμε κοινό αγώνα για δράση ώστε στο μέλλον να έχουν όλοι μια καλύτερη ζωή. Εγώ ασχολούμαι με τον πολιτισμό με νέους εδώ και 30 χρόνια και με πτωχότερους πολίτες και ξέρω ότι η διαμεθοριακή συνεργασία πέρα από φραγμούς και σύνορα δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν οι νέοι ότι οι προσπάθειές τους έχουν αποτέλεσμα. Στο βορρά της Γερμανίας υπάρχει ένα σχολείο ειρήνης όπως λέγεται που ιδρύθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οι καλλιτέχνες που εργάζονται εκεί συμπεριλαμβάνουν και μερικούς Βρετανούς, έναν Βρετανό που γνωρίζω που κάθε καλοκαίρι πηγαίνει και φέρνει πληροφορίες και δραστηριότητες πολιτιστικές για όλους τους νέους που έρχονται εκεί. Οι νέοι που συμμετέχουν προέρχονται από πολλά κοινωνικά στρώματα και χώρες. Θα μπορούσε κανείς να νομίσει ότι έχουν ρετσιστικές απόψεις για τους άλλους λαούς, αλλά όχι. Όχι. Μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους γνωρίζοντας άλλους. Μαθαίνουν να ε, είναι και πιο επιτυχείς, πιο αισιόδοξοι και οι νέοι με τους οποίους έχω συνεργαστεί εγώ για τόσα χρόνια, μερικούς τους γνωρίζω από μικρούς, τώρα είναι 20-30 χρονών, είναι εκείνοι που είναι οι πιο πετυχημένοι στην κοινότητά μου. Μαθαίνουν να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και έτσι να επαναφέρουν την οικονομική ανάπτυξη στις κοινότητές τους. Είναι λοιπόν αναλυθεί όλα όσα είπε η κυρία Λουίζα. Εξάλλου και στο Στρασβούργο ντράπηκα όταν είδα πως δρούσε το UKIP. Ντρέπομαι που έχουμε την ίδια εθνικότητα και δεν πρέπει να νομίζετε ότι οι περισσότεροι Βρετανοί πρεσβεύουν τα του UKIP. Στα βορειοδυτικά της Αγγλίας οι περισσότεροι εκλογείς θέλησαν εργατική διοίκηση και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι στο Μάντσεστερ είναι από το εργατικό κόμμα και υποστηρίζουν πολιτιστικά προγράμματα όπως το να γίνει το Birmingham πόλη πολιτισμού. Και αυτό είναι ουσιώδες. Όχι μόνο για τον βρετανικό πολιτισμό αλλά διεθνώς για τον ευρωπαϊκό. Ο κύριος Φαράτζ είπε, ο Νάιτζελ Φαράτζ, ότι αισθάνεται ότι τον μισούν στην Ευρώπη. Θα ήθελα να του πω να έρθει μαζί μας και να δει τι κάνουμε πολιτιστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να δει πώς θα μπορούσε να αγαπηθεί από την Ευρώπη αντί να τον μισούν όλοι. Εγώ στις κοινότητες που δρώ ξέρω ότι είναι όλοι αγαπητοί γιατί πιστεύουν ότι η πολιτιστική συνεργασία και η τέχνη είναι καλύτερος τρόπος για να έχουμε ένα κοινό μέλλον αντί να στρέφουμε τα νότα στους γείτονές μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τα τόσα συνεπρακτικά μας είπατε. Και τώρα, ο κύριος Εύανς έχει το λόγο. Η κυρία Εύανς. Um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι νέο ευρωβουλευτή, αλλά είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή μας και περιμένω πώς και πώς για όλα τα ενδιαφέροντα που θα κάνουμε. Προέρχομαι από την Ουαλία, τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είμαστε δίγλωση περιφέρεια της χώρας και είμαστε υπερήφανοι για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Επίσης, έχουμε αναπτύξει την βιομηχανία στην περιφερειά μας και η Ευρώπη θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για τον κλάδο αυτό. Η οικονομία μας έχει μετασχηματιστεί, ε, βεβαίως και πάρα πολλούς καλλιτέχνες έχουμε, οι οποίοι ενατενίζουν την προσπάθεια για βοήθεια προς αυτούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και το Erasmus Plus είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλοί νέοι μέσω του έρασμος έχουν έρθει εδώ στις Βρυξέλλες. Άλλαξε η ζωή τους έτσι. Τους ξενύχθηκαν νέες ευκαιρίες. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαντικό πρόβλημα είναι η ανεργία των νέων, αλλά μπορούμε έτσι να δώσουμε στους νέους κάποιες φρέσκες εμπειρίες και ένα καλύτερο μέλλον. Ευρώπη σημαίνει πολυμορφία. Σημαίνει πολλές γλώσσες, σημαίνει μειονοτικές γλώσσες. Και στα μέσα ενημέρωση και το θέμα είναι πώς εμείς θα βοηθήσουμε όλους ούτω ώστε να μπορέσουν να βρίσκονται κοντά στην ταυτότητά τους κλπ. Και ο αθλητισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, είναι κάτι όλο ένα και πιο σημαντικό. Και συμφωνώ με τις προτάσεις που έκανες, Πρόεδρε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε, κυρία Εύανς. Ο κύριος Γραμματικά έχει το λόγο. Χαίρομαι πολύ για την ε, σημερινή πρώτη συνεδρίαση και είμαι βέβαιος ότι με την Προεδρία σας, κυρία Πρόεδρος, και την εμπειρία σας ε, αυτή η Επιτροπή πολύ σημαντική του πολιτισμού και της παιδείας ε, θα χαράξει έτσι πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές. Και πρέπει να πω ότι επειδή σε αυτή την Επιτροπή ακούστηκαν απαράδεκτες θα έλεγα εκφράσεις εναντίον του πολιτισμού και είναι πρωτοφανές άνθρωποι να συμμετέχουν σε μια επιτροπή και να καταγγέλουν το ρόλο της ίδιας της επιτροπής. Διερωτάται κανείς τι κάνουν εδώ μέσα. Υπάρχουν αλλού ίσως ε, ευήκοα αυτιά, πολύ λίγα νομίζω, για να ακούσουν τα όσα λένε. Θα προχωρήσω στο δυσάρεστο γεγονός που μου αναφέρατε ότι υπάρχουν περικοπές ε, νομίζω πρέπει να γίνει οτιδήποτε δυνατόν. Δεν έχω πλήρη εικόνα του προϋπολογισμού, αλλά πρέπει να σας τονίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι ο πολιτισμός, ειδικά στις χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, μια από τις οποίες ίσως και η πιο οδυνηρή είναι στην Ελλάδα, ο πολιτισμός είναι μια ανάσα. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, Ξέρω ότι όλα τα προγράμματα, τα Erasmus, τα Erasmus Plus, πόσο πολύτιμα είναι για τους ε, φοιτητές μας, για τους σπουδαστές μας και ελπίζω να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να κερδιθούν, όχι να χάσουμε ποσά, να κερδίσουμε ποσά από το γενικό προϋπολογισμό. Θέλω να είμαι αισιόδοξο, γιατί και εμπειρία υπάρχει και θέληση. Και να τελειώσω με μία παρατήρηση. Η χώρα η δική μου, η Ελλάδα, δεν έχει μόνο καθιερωμένες ε, αξίες στον πολιτισμό, όπως είναι η λυρική σκηνή, το εθνικό θέατρο, ο Μίκης Θεοδωράκης, ε, τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες. Έχει και νέους ανθρώπους, πάρα πολύ σημαντικούς, νέες ομάδες καλλιτεχνών, ε, που ήδη έχουν δώσει λαμπρά δείγματα στον κινηματογράφο, στην τέχνη και αυτοί πραγματικά προσβλέπουν προς την Ευρώπη θα έλεγα για μια χείρα βοηθείας που δεν είναι πάντα οικονομική, είναι ένα ενδιαφέρον, είναι μια μέρημνα ε, για να ανοίξουν αυτό το δρόμο που τόσο προσδοκάμε. Και βέβαια στην παρατήρηση του συναδέλφου μου του κυρίου Γλέζου για τα τοπονύμια νομίζω της Κύπρου ότι έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω και να πω ότι οι τοπικές ιστορίες πρέπει να είναι σεβαστές όσο είναι δυνατόν και κλείνω και πάλι με κάποια αισιοδοξία. Υπό την Προεδρία σας νομίζω ότι θα ανοίξουμε και νέους δρόμους σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική για τις μέρες που ζούμε επιτροπή. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Γραμματικά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις ευχές σας την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είμαι νέο μέλος και ίσως βέβαια επειδή δεν γνωρίζω τα πράγματα ακόμη να κάνω και κάποια λάθη σε αυτά που θα πω αλλά ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά. Ελπίζω ότι και η Πρόεδρος και όλοι μας θα πράξουμε πάντο δυνατό για να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής μας. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός, η παιδεία, η εκπαίδευση θα βοηθήσουν την Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση. Εγώ είμαι και φοιτήτρια, είμαι και καθηγήτρια. Και έχω την ευκαιρία να δω πόσο σημαντικές είναι οι ανταλλαγές των σπουδαστών. Αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων θα παρακαλέσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτισμού να διαθέσει περισσότερα έγγραφα στους βουλευτές, ιδίως στους νέους βουλευτές. Για παράδειγμα, τον προϋπολογισμό προηγούμενων προγραμμάτων, που δεν έχουμε γνώση και θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Αντινόρφη. Κύριος ή κυρία Ζαμπάσκη. Θα μιλήσω βουλγαρικά, κύριε Πρόεδρε. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μένω κάπως έκπληκτος διότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού πάει να γίνει σύγκρουση μεταξύ κομμάτων και σύγκρουση ιδίως μεταξύ βρετανικών κομμάτων. Παρακαλώ όλες και όλους να δείξετε σεβασμό απέναντι στις απόψεις των άλλων. δεν ενδιαφέρει τόσο η γνώμη του ενός κόμματος και του άλλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η φωνή των πολιτών. Αυτήν μεταφέρουμε εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ακούσουν όλους και όλες. Καθένας είναι σημαντικός εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων στον χώρο του πολιτισμού, ασφαλώς και είναι σημαντικό να υποστηριχθούν από την, Ευρωπα... από την ε, Επιτροπή μας. Για μένα και του συναδέλφους μου είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία των προγραμμάτων, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την ιδιαιτερότητα ή τι ιδιαιτερότητε τη κάθε μια χώρα μέλου. Γιατί κάθε χώρα μέλο έχει τα δικά τη χαρακτηριστικά, τι ιδιαιτερότητέ τη. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια ενισχυμένη χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Αυτή η ενισχυμένη χρηματοδότηση θα πρέπει να επιτρέψει να γνωρίσουμε και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας χώρας. Είναι διαφορετικό αν ζει κανείς στο Ιράν ή στην Κύπρο ή στην Πορτογαλία. Κάθε χώρα είναι υπερήφανη για τον πολιτισμό της, για τη γλώσσα της και ούτω καθεξής. Και είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την πατρίδα μου. Σας εύχομαι λοιπόν καλή δουλειά σε όλες και όλους στην, μέσα στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε βέβαια στα λόγια, αλλά σε πραγματικό αμοιβαίο σεβασμό. Σόιντρόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι από τα καινούρια μέλη στην Επιτροπή αυτή. Και επειδή φαίνεται ότι όλοι ζητούμε να υποστηρίξουμε την πολυγλωσία, θα μιλήσω και εγώ στην ωραία μου μητρική γλώσσα. Ένα από τα βασικότερα προγράμματα που στηρίζει ο Έρασμος είναι το πρόγραμμα Comenius, που είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε πολύ. Έχουν γραφτεί πολλοί φοιτητέ στο πρόγραμμα αυτό που ονοματίζεται από την προσωπικότητα του Τζον Έιμς Κομίνιος που προέρχεται από την περιφέρειά μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ιδέες που εξέφρασαν για τη βελτίωση του προϋπολογισμού του 2015 και στηρίζω ιδιαίτερα την τροπολογία του κυρίου Στογεύσκη για τις εταιρικές σχέσεις με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα με την Ουκρανία. Πιστεύω ότι οι χώρες που μετά το κομμουνιστικό τους παρελθόν κινήθηκαν προς τη δημοκρατία είναι σημαντικό να στηριχθούν μέσω της παιδείας και αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει από την Ένωση. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτήν την ε, τροπολογία. Πρέπει να δούμε όμως και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ποσά αυτά. Η τσεχική δημοκρατία αποφάσισε να υποστηρίξει την Ουκρανία με πολλά εκατομμύρια κορώνες μέσω ιδιωτικών ομίλων και οργανισμών, οργανώσεων. Ελπίζω όλοι να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία και θα ήθελα οι συνάδελφοι που δεν είναι ικανοποιημένοι για με τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή ιδίως από μία συγκεκριμένη χώρα πρέπει να καταλάβουν ότι η παιδεία είναι τμήμα του, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δική μου εκλογή αυτό αναμένουν από μένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ, στα γερμανικά αυτή τη φορά. Επανέρχομαι σε αυτήν τη διαμάχη που παρακολουθήσαμε πριν. Ο εθνικισμός αλλά και ο υπερτονισμός του εθνικισμού γνωρίζουμε που οδήγησε στον προηγούμενο αιώνα. Κατέστρεψε την Ευρώπη. Οπουδήποτε αναφύεται ο εθνικισμός βλέπουμε ότι δεν λύνει κανένα πρόβλημα, μόνο προκαλεί νέα. Και γι' αυτό αν δει κανεί την επιτυχία των διασυνοριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τους σπουδαστέ, για τα σχολιά που συνεργάζονται, για μικρά παιδιά τα οποία έρχονται σε επαφή με άλλους συμμαθητές τους από άλλα σχολιά, από άλλες χώρες. Βλέπουμε τι μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Δίνουν στους πολίτες της Ευρώπης κοινού σκοπούς, χωρίς να υπερέχει μια χώρα απέναντι στην άλλη. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Και αν ρίξει κανείς απ' έξω μια ματιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπει πόσοι άνθρωποι θεωρούν ότι αξίζουν τα προγράμματα αυτά. Αυτά θέλω να υπενθυμίσω και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης χρηματοδότηση των προγραμμάτων και θα αγωνιστούμε για αυτήν. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με υπερεθνικιστικές κορώνες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία παρέμβαση από την Αντιπρόεδρο κυρία Μπόξορ. I uh, Ας μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, τα Ουγγρικά. Πρώτα πρώτα. Να επανέλθω σε κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Δηλαδή να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός. Ήδη είδαμε κατά αυτόν τον αιώνα και όχι μόνο πόσο ο πολιτισμός βοήθησε την διπλωματία. Πώς είχαμε ανακοχή, ειρήνη, ε, πέρα των, των, των πολέμων χρησιμοποιώντας την συνεννόηση, την διαπολιτισμική. Έτσι βοηθήθηκε και η ανάπτυξη, έτσι τελικά πετύχαμε κάποια εξέλιξη σε όλα. Οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τα προγράμματα ανταλλαγής στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Είναι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν να γνωρίσουν τον κόσμο, να δουλέψουν σε ξένες χώρες. Και έτσι αποκτούν ένα πλεονέκτημα για να ενταχθούν έτσι καλύτερα στον κόσμο της δουλειάς. Θα πρέπει πάνω σε αυτά να διαμορφωθεί συνένεση. Ή βέβαια υπάρχει και η UNESCO η οποία βοηθά. Έχουμε τις ε, έρευνες που γίνονται και για τη γεωργία και για αλλού. Εκεί όπου τα πράγματα γίνονται δύσκολα λόγω ε, συγκρούσεων που εκεί σώβουν. Θα πρέπει επίσης αυτά τα προγράμματα να επεκταθούν και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και έτσι θα πετύχουμε προσέγγιση των λαών. Ουκρανία. Mm. Τα έχω πει και επαναλάβει. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει την επιθετικότητα όπως εκφράστηκε εκεί. Και από τις δύο πλευρές βέβαια, αλλά κυρίως από πλευράς των αυτονομιστών. Θα πρέπει επίσης να παράσχουμε βοήθεια με τα προγράμματα εταιρικής σχέσης που υπάρχουν, έτσι να πλαισιώσουμε την Ουκρανία και να έχουμε επίσης και προγράμματα ανταλλαγής με τη χώρα εκείνη. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπόξορ. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και από πολιτικής και πολιτιστικής πλευράς. Κάποιες σκέψεις μου τώρα. Είναι σωστό να σεβόμαστε όλους τους αδέλφους όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όλοι συμμεριζόμαστε την αξία της ύλη της επιτροπή μας. Ξέρουμε με θέματα νεότητας, με θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και όλοι έχουμε χωνέψει το ότι εάν δεν μπορούμε να έχουμε βελτίωση ποιοτική με κάποιους προγράμματα διασυνοριακά σε αυτά στα πολιτιστικά και επιστημονική για τους νέους αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ειρηνική ύπαρξη. Αυτό γίνεται μέσω της γνώσης του άλλου, μέσω του αλληλοσεβασμού, όπως τα είπε η κυρία Μπόξορ, γνώση της ιστορίας. Έτσι είναι σε όλες τις συγκρούσεις και σε όλες τις αντιπαραθέσεις. Έχει επομένω διπλή υφή και σχέση ο πολιτισμός ότι δηλαδή αναπτύσσεται και το άτομο αλλά και έτσι έχουμε καλύτερη κοινωνική συνοχή. Αυτό βοηθάει και την ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία. Έτσι θα πρέπει να διαμορφώνουμε τις τοποθετήσεις μας. Τώρα, θελήσατε ενημέρωση σε κάποια ζητήματα. Είπαμε ότι είναι στη διάθεσή μας ε, η γραμματεία, μπορεί να σας ενημερώσει αυτά που ζητήσατε και για τα ποσά και για τις ακροάσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό, σε σχέση με τα όσα έχει προτείνει η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Κυρία Ερθαβάλα Ρουμπιάλ είναι ε, η είναι αν τρία εδώ στην Επιτροπή μας έχει αναφέρει την εισήγηση για όλο το Κοινοβούλιο και θα συνεργαστούμε μαζί που είναι πολύ σημαντικό και επίσης οι τροπολογίες που θα προτείνω κατά συνεννόηση με τις άλλες επιτροπές και θα ψηφίσουμε τον ε, Σεπτέμβριο αφού συνηθούμε και με τους σκιώδεις ηγητές. Έτσι θα προστατεύσουμε, θα αυξήσουμε τον προπολογισμό και εγώ με μεγαλύτερη επιμονή, όπως σας είπα στην αρχή, θα προσπαθήσω να πω το ότι οι περικοπές στο τρίτο κεφάλαιο για αυτό το 3,3% ε, που αφορά τα προγράμματά μας θεωρούμε ότι δεν είναι συνεπές σε σχέση με αυτά τα οποία θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και εν ώψη της στατικής για το 2020. Όσοι εισηγήτρια, σας το υπόσχομαι. Και είμαι βέβαιη ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων στην Επιτροπή μας θα είναι μαζί μου. Τώρα έχουμε την κυρία Μπριζίτ ε, εγώ από την Γενική Διεύθυνση για τα Πολιτιστικά που θα μας μιλήσει, Προεδράς Επιτροπή και κατόπιν Γιάννη από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Ε, ποιος θα λάβει το λόγο, ποια από τις δύο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και τις συστάσεις σας και την υποστήριξη για τα πολιτιστικά προγράμματα. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικά σχόλια για το MFF και την κατάσταση του προϋπολογισμού το 14 και πώς θα επηρεάσει το 2015. Είναι βέβαια πολύ πιο τεχνικό αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες. πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποφασίστηκε από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2015. Το έρασμα ΣΥΝ έχει αυξηθεί κατά 14% για την αύξηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα. τα τελευταία τρία χρόνια του Πολδίπ, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι τα σημαντικότερα. Για τις μαθητείες των νέων ιδιαίτερα υπήρξε χρήσιμο το έρασμος συν για καλύτερη και περισσότερη απασχολησιμότητα, για περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της Ευρώπης. Για το Creative Europe το Πολδίπ προτείνει 19% αύξηση από το 16 μέχρι το 19 δηλαδή ετήσια αύξηση περίπου 15% και ακόμη 5% το χρόνο μέχρι το 20. Το 14 και τις αρχές του 15 προτείνονται μικρές αρχικές περικοπές αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις ως προς τις δανειοδοτήσεις ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών οικονομικών τομέων. Επειδή υπήρξαν λοιπόν το 14 ορισμένες μικρές περικοπές, η Επιτροπή Πολιτισμού πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού για το Creative Europe και τελικά πήρε 2 δισεκατομμύρια παραπάνω. On Για τις πληρωμές έχουμε πολύ μεγάλη πίεση για τις οροφές των κοντιλίων που προβλέπει το Πολδίπ. Τα επίπεδα προχρηματοδότησης βρίσκονται στο, στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο στάδιο και αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ροή στους συμμετέχοντες. Επειδή λοιπόν ήδη από το 11 και 13, τους του 11 με 13, είχαμε πολύ μεγάλη πίεση για τις πληρωμές, ο προϋπολογισμός του 14 είχε χαμηλά κονδύλια για τις πληρωμές, ας πούμε για το έρασμος συν, χρειάστηκε η μείωση της προχρηματοδότησης αλλά για να ε, υπάρξει, να συνεχιστεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος οι περικοπές ήταν περιορισμένες εφόσον μάλιστα πρόκειται για σχολεία και φοιτητές που δεν έχουν τα έσοδα με τα οποία να περικόψουμε παραπάνω την προχρηματοδότηση. Την περικόψαμε όσο μπορούσαμε αλλά όχι υπερβολικά. Τα 2 εκατομμύρια όμως δολάρια πληρωμών για φέτος προβλέφθηκαν από τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2014 και τώρα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τα δε 202 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα ανταλλαγών Da στα πλαίσια του Εράσμου για το 14 και 15. Ευτυχώς για το Creative Europe δεν χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα για μείωση της προχρηματοδότησης. Για το 2015 τώρα η Κομισιόν πρότεινε για τις προβλέψεις να ακολουθήσουμε ό,τι πρόβλεπε το Πολδίπ. 14% αύξηση δηλαδή για το Erasmus Sin και 9% για το Creative Europe σε 7 ετή περίοδο. 2,1% αύξηση δηλαδή για το Erasmus. 2. Είναι ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή νομίζω. Χρηματοδοτούμε 208.000 φοιτητές, 280.000 φοιτητές περίπου στα πλαίσια του Λεωνάρδο Νταβίντσι και για το πρόγραμμα Youth in Action χρηματοδοτούμε τις ανταλλαγές μεταξύ 76.000 νέων. Όλα αυτά θα βοηθήσουν για την πραγματοποίηση των στόχων που εξηγήσατε όλοι σας πριν. Επίσης έχουμε το δημοσιονομικό μέσο της δανειοδότησης φοιτητών που ωφελεί 13.000 φοιτητές μάστερς. Υπάρχει και η εξωτερική διάσταση του έρασμος συν που θα επιτρέψει σε πάνω από 20.000 φοιτητές να έρθουν στην Ευρώπη για να σπουδάσουν, ιδιαίτερα από την Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Yes. Then, regarding the... Και για τις πληρωμές για το 15 του Ερασμοσίν, δεν είχαμε πολλές δυνατότητες για τις πληρωμές διότι και γι' αυτό η Κομισιόν έβαλε τα κατώτατα ποσά που απαιτούνται για να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα το 2015. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ξαναεφαρμόσουμε το μέτρο που ονομάζεται μείωση του ελλείμματος, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ξαναχρειαστεί διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2015. Τώρα για το Creative Europe Υπάρχουν μικρές περικοπές 1,7% στις προβλέψεις. Η Κομισιόν πρότεινε να μειωθούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα και για, το, για μικρά προγράμματα όπως τηλεοπτικά, κινηματογραφικά κλπ. Παρόλα αυτά, θα ενισχύσουμε στα πλαίσια του ίδιου εργαλείου τα τεχνικά προγράμματα και μέτρα που να διευκολύνουν στους δημοσιονομικούς ενδιαμέσους να ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα αυτό και να αρχίσουν από το 16 τουλάχιστον να εφαρμόσουν τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον πολιτιστικό τομέα. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μικρές περικοπές που προβλέπονται για το 2015 για το Creative Europe είναι οι μάξιμου περικοπές που μπορούσαμε να κάνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι οποιασδήποτε περαιτέρω περικοπές θα πρέπει να αποφασιστούν από την διαδικασία έγκρισης του προπολογισμού, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι καταστροφικές για το πρόγραμμα και για τον πολιτιστικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δρούν στα πλαίσια του. Επίσης, το 2015 δεν θα λειτουργήσει το Ταμείο Εγγυήσεων, δεν θα λειτουργήσει Ταμείο Εγγυήσεων και γι' αυτό το Creative Europe πρέπει τουλάχιστον να έχει τα ποσά που προτείνει η Κομισιόν. Uh, Τώρα να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που ακούστηκαν. Το πρώτο αφορούσε την μη φορολόγηση των προγραμμάτων του Έρασμος συν οι δαπάνες της Κομισιόν εφαρμόζονται με αυστηρούς κανόνες που είναι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί και θα εξετάσω τα πράγματα και θα μπορέσω να σας απαντήσω γραπτός λεπτομερέστερα για τις διαφορές μεταξύ χωρών μελών και τις αποκεντρωμένες δράσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κονδύλια το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Έρασμου ΣΥΝ και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών δημοσιεύονται στο ίντερνετ. Για το 2015 δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τα κράτη-μέλη τα ποσά. Είναι πιθανό η Κομισιόν μέσα Αυγούστου, 15 Αυγούστου να το εγκρίνει. Και θα το βρείτε στο ίντερνετ ε, υπό τον τίτλο «Ο Ιρώπα. για τα αθλητικά προγράμματα ένας από τους στόχους του ΕΡΑΣΜΟΣ Συν είναι ο υγιής τρόπος ζωής. Τα αθλητικά προγράμματα είναι κάτι το καινούριο από το 14 μόνο και μετά. Ο προϋπολογισμός τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια αλλά επειδή είναι καινούριο, κάτι καινούριο θα αρχίσει με χαμηλά ποσά και μετά θα αυξηθούν όταν αρχίσουν ήδη να εφαρμόζονται τα πρώτα προγράμματα. Τα συγκεκριμένα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν στον αθλητικό τομέα επίσης θα τα βρείτε στο πρόγραμμα εργασιών του Erasmus συν στο ίντερνετ. Uh, Για την Ευρωπαϊκή η Εβδομάδα Κινηματογράφου το 14 το προϋπολογισμό τους τον είχαμε βάλει σε μια χωριστή θέση του προϋπολογισμού, του γενικού προϋπολογισμού, αλλά βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού εφόσον υπάρξει νομικό υπόβαθρο πρέπει οι δραστηριότητες να εφαρμοστούν σύμφωνα με αυτό. Άρα οι προβλέψεις για τα αθλητικά του Έρασμος 2 και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινηματογράφου καθώς και τον... Αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο τομείς πρέπει να αποφασιστούν μετά από διαγωνισμούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε χρήματα εάν ένα πρόγραμμα δεν προβλέπεται από το νομικό υπόβαθρο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινηματογράφου πήρε το εκατομμύριο που ζητούσε γιατί το ενέκρινε και η Κομισιόν και νομίζω αυτά είχα να σας πω. Ε, ε σας ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Ντεβόστ, για την πολύ λεπτομερή απάντηση που δώσατε στα σχόλια των συναδέλφων μου. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να παρέμβουν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί είστε η κυρία Ντούρκοβιτ. Ευχαριστώ κυρία Πάρα. Είναι περιορισμένος ο προϋπολογισμός των επικοινωνιών. Ωστόσο έχει ως χρέος να ενημερώνει 500 και εκατομμύρια πολίτες. Ενώ έχουμε 243 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις υποχρώσεων, ανάληψη υποχρώσεων. Λίγο αυξημένο σε σχέση με το 2014 και 23 εκατομμύρια παραπάνω από το 2013. Χωρίζουμε τον προϋπολογισμό μας σε τρία κεφάλαια. Πρώτον, διοικητικές δαπάνες που καλύπτουν και τις δαπάνες της έδρας αλλά και των εκπροσωπήσεών μας. Δεύτερο, η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και το πρόγραμμα Ευρώπη για τον πολίτη. Και το τρίτο μέρος βεβαίως βασίζεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό του 2014, μειώθηκε όμως για φέτος κατά 1,1 εκατομμύριο απέναντι στο προϋπολογισμό του 2014 και περίπου 3 απέναντι στο προϋπολογισμό του 2013 και θα γίνουν και άλλες περικοπές από το Συμβούλιο. Ένα εκατομμύριο στις υποχρώσεις και άλλο ένα στις πληρωμές. Ελπίζουμε να μας χορηγήσετε την υποστήριξή σας για να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον, αν δεν έχουμε δηλαδή αύξηση, τουλάχιστον να αποκαταστήσουμε το ποσό που έχει προβλέψει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προπολογισμό. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο προβλέπει τις καθ' αυτό επικοινωνιακές δράσεις. Έχουμε αύξηση απέναντι στο προϋπολογισμό του 13 κατά 13 εκατομμύρια και απέναντι στο προϋπολογισμό του 14 κατά 4 εκατομμύρια φέτος. Πιο πολλοί βέβαια έχουν μειώσει κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ τις πιστώσεις πληρωμών. Αυτά βέβαια είναι και προνόμια του Συμβουλίου. Όμως οι πιστώσεις πληρωμών είναι κέρια σημασίας για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Το 2013 είχαμε 5,8 εκατομμύρια στις πιστώσεις πληρωμών, όμως δεν έγινε δεκτή η αύξηση αυτή και επομένως ο προϋπολογισμός του 2014 χρειάστηκε να καλύψει τα ποσά από το 2013. Για τα κενά του 2014 θα χρειαστούμε πάλι ενίσχυση των πιστώσεων στα πλαίσια μιας συνολικής μεταφοράς πιστώσεων. Ιδεμή δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις πληρωμές, να πληρώσουμε δηλαδή όλα όσα χρωστάμε με άλλα λόγια η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή, ή μάλλον δική σας Επιτροπή, να επανέλθει στα αρχικά ποσά του σχεδίου προπολογισμού της Ένωσης για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές, εμάς μας ικανοποιεί αυτό και αν ακόμα προβλέψετε αύξηση του προγράμματος η Ευρώπη υπέρ του πολίτη, θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένες αν καταφέρετε να αυξήσετε κατά ένα εκατομμύριο τις πληρωμές. Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών σας ενημερώνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει πιστώσεις για το Evranet. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να ανανεώσουμε τη σύμβαση για την Ευρανέτ στο τέλος του 2015 εκτός εάν βρεθούν χρήματα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου για την πολύ ε, λεπτομερή περιγραφή της καταστάσεως. Σίγουρα η Επιτροπή Πολιτισμού θα υποστηρίξει τα αιτήματά σας που δεν είναι αίτημα μοναχά της Γενικής σας Διευθύνσεως αλλά είναι κοινό αίτημα γιατί γνωρίζουμε τη σημασία των προγραμμάτων αυτών και βεβαίως σε μια περίπτωση όπου ακόμα δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες και δεν ενημερώνονται αρκετά οι πολίτες για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα νέα προγράμματα. Βρισκόμαστε σε μια φάση δηλαδή όπου καλούμεθα να εξηγήσουμε στους πολίτες τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Άρα οι δραστηριότητες επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτά που μας λέτε λοιπόν ασφαλώς ανταποκρίνονται και στις δικές μας προσδοκίες και ως Επιτροπή Πολιτισμού θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή για τον προπολογισμό. Βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Μιλήσαμε και για πιλωτικά προγράμματα και για προπαρασκευαστικές δράσεις και πολλούς από εσά σας ενδιαφέρουν αυτά. τέλος Ιουλίου είναι η προθεσμία για να υποβληθούν τα πιλωτικά προγράμματα. Βέβαια, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια από αυτά απέδωσαν και ποια όχι. Όμως, τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία ήδη έχουν λειτουργήσει θα πρέπει να τα περιλάβετε σε τροπολογίες στον προπολογισμό. Ορισμένοι από εσάς ήδη τα θίξατε αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η ανατολική γειτονία, η συνεργασία δηλαδή με τους ανατολικούς γείτονες. Υπάρχει και το πρόγραμμα Erasmus Mundus που έχει τον ίδιο στόχο. Επίσης η Δημιουργική Ευρώπη, Europe Creative, η Creative Europe. Επίσης αυτές, αυτά τα προγράμματα απευθύνονται και σε τρίτες χώρες. Δίνουν λοιπόν μια ευρεία εικόνα της Ευρώπης. Έχουν μάλλον ένα ευρύ όραμα για την Ευρώπη τα προγράμματα αυτά ευρύτερο από την Ένωση. Η προθεσμία όμως υποβολής τροπολογιών λύγει αύριο το μεσημέρι για τροπολογίες που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα νούμερα. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε το προϋπολισμό και στα κείμενά του δηλαδή και στα σχόλια αλλά και για τα ποσά, τα συγκεκριμένα ποσά. Πριν από τις 4 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει αυτό, ίσως στις 2 Σεπτεμβρίου. Θα αποφασίσουμε από κοινού πότε θα γίνει η συνεδρίαση αυτή και ενδεχομένως θα χρειαστεί να αναζητήσουμε και συμβιβασμούς. Να συγχωνεύσουμε δηλαδή τροπολογίες που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο έτσι ώστε να συναποτελέσουν συμβιβαστικές τροπολογίες. Αν ίσως έχετε ερωτήσεις τώρα ή άλλα θέματα να θίξετε, έχει καλό να το πράξετε τώρα, αλλιώς θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη των προσεχών συνεδριάσεων. 3 και 4 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, 4 Σεπτεμβρίου το πρωί και θα είναι βεβαίως ήδη υπό Ιταλική Προεδρία. Άρα η αντίστοιχη Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού θα είναι παρόντες και στις 4 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, θα ψηφίσουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού και τα κείμενα των τροπολογιών. Και αν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, τότε μπορούμε ίσως να κάνουμε μια παρουσίαση του τμήματος μελετών του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Γλέζος ζήτησε να ενημερωθεί περισσότερο για τις μελέτες που υλοποιούνται καθώς επίσης και για τις αποστολές που μπορεί να αναθέσει κανείς στο τμήμα μελετών. Επίσης, εκπρόσωπος της Γενικής Διευθύνσεως Πολιτισμού θα είναι παρόν. Αν προλαβαίνουμε λοιπόν θα τα κάνουμε αυτά στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα, θα μπορέσουμε τότε να γνωρίσουμε και τον νέο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτισμού. Θα μας επιτρέψει αυτό να έχουμε καλύτερη εικόνα τότε των μελετών που μπορεί να ζητήσει κανείς από το τμήμα μελετών. Αυτά. Αν δεν έχετε άλλο τίποτε στα διάφορα, τότε νομίζω μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στη συζήτηση. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και νομίζω ότι μετά από τον δύσκολο εκλογικό αγώνα όλοι έχουμε ανάγκη από διακοπές. Σας ευχαριστώ.